Καθυστέρησα λίγο την έναρξη της συνάντησης, γιατί ίσως κάποιοι από εμά ασχολήθηκαν περισσότερο με τους αγώνες του ποδοσφαίρου που τελειώνουν όπου να είναι και θα έρθουν μαζί μας σε λίγο. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους σήμερα. για μια συνάντηση την οποία θα αφιερώσουμε σχεδόν ολοκληρωτικά στις σχέσεις της Ένωσης με τον ΝΑΤΟ. Να σας θυμίσω ότι έχουμε αρκετές γλώσσες στη διάθεσή μας. Λέει τις γλώσσες ο πρόεδρος οι οποίες δεν θα ακούγονται σήμερα. Ταυτόχρονα μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη την κάνουμε δεκτή. Να σας θυμίσω ότι στις 17 Ιουνίου το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την Ισραηλινή ενέργεια κατά της ανθρωπιστικής, του ανθρωπιστικού στολίσκου. Ζητήθηκε από την ΥΠΑ το εκπρόσωπο να επανεξετάσει την εντολή της ε, αποστολής βοήθειας και γι' αυτό θα οργανώσουμε σύντομα μία συνάντηση για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή. Ξέρετε ότι υπάρχει αποστολή και στη Ράφα και σε άλλα μέρη. Μετά τις διακοπές θα συζητήσουμε τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της ασφάλειας στην Αφρική, ιδιαίτερα στη Γουινέα Μπισάου και στην Δημοκρατία του Κονγκό. Θα κάνουμε γενικά ένα, θα έλεγα, μια συνολική συζήτηση για θέματα αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές της Αφρικής αλλά και στη Γεωργία. Περιμένω και κάποιους Βούλγαρους συναδέλφους σήμερα από την Βουλή της Σόφια. Αν είναι εδώ τους καλωσορίζω. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τον Τζέιμι Σέι, τον ξέρετε όλοι. Είναι διευθυντής προγραμματισμού και τέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Το Ζων Φρανσουά Μπυρό δεύτερος γενικός γραμματέας για τη δημόσια διπλωματία και δύο μονίμους εκπροσώπους. Το Πολωνό εκπρόσωπο στο ΝΑΤΟ και την κυρία Ανδρεανή, μόνιμη εκπρόσωπο της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ που βρήκατε χρόνο να έρθετε εδώ σήμερα. Στόχος είναι να δούμε την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υπό την καθοδήγηση της κυρίας Όλμπραιτ και υπό το φως της εκθέσεως αυτής να συζητήσουμε τις νέες αντιλήψεις για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το ΝΑΤΟ. Και να μιλήσουμε επίσης πιο ειδικά για τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, που συζητήθηκε τη Δευτέρα γιατί ο Γενικός Γραμματέας Ράσμουσεν ζήτησε να υπάρξει μια εταιρική σχέση στρατηγικού τύπου ανάμεσα στην Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θα συναντηθεί ο πρόεδρος Μπούζεκ με τον Ράσμουσεν τον Ιούλιο και μετά από τη συνάντηση στη Ρίγα, στη Ρίγα την κοινοβουλευτική και πήρε ε, μέρος ο κύριος Σαρουσβόλσκι που μόλις μπαίνει στην αίθουσα. Υπήρξε μια πρόκληση προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να έρθει να πάρει το λόγο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη δική μας υποεπιτροπή. Τα θέματα λοιπόν τρέχουν, πολλά ερωτηματικά τίθενται, και θα ήμουν ευγνώμων από τους προσκεκλημένους μας σήμερα να μας μεταφέρουν τις αναλύσεις τους και να εμπλουτίσουν τη συζήτηση αυτή. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον πρέσβη της Πολωνίας, μετά στην κυρία Ανδρεάνη και μετά στον κύριο Οσί και μετά στον Πυρό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συναντούμε εδώ σήμερα. Η συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ένωση έχει πολύ μεγάλη σημασία και την εκτιμούμε δεόντως. Να ξεκινήσω με κάποια λόγια για τις διαδικασίες, πώς δηλαδή αναπτύσσεται η στρατηγική αντίληψη και ποιες είναι οι βασικές αρχές με τις οποίες λειτουργήσε η ομάδα των εμπειρογνωμόνων και πώς αυτό εντάσσεται στη σύνολη διαδικασία. Βασική ιδέα αυτής της προσπάθειας ήταν η μέγιστη διαφάνεια και η συλλογή της εμπειρογνωμοσύνης από πάρα πολλές πλευρές και βλέμματα. Νομίζω ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ, η διαβούλευση ή το ευρυτάτη. Να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε τέσσερα στρατηγικά σεμινάρια στο Λουξεμβούργο, τη Λιουμπλιάνα, το Όσλο και τη Βόσινγκτον. Σε κάθε ένα από αυτά τα σεμινάρια ασχοληθήκαμε με συγκεκριμένα θέματα τους βασικούς λόγους της συμμαχίας στο Λουξεμβούργο, συνολική αντιμετώπιση στη Λιουμπλιάνα, εταιρικές σχέσεις στο Όσλο και το τελευταίο σεμινάριο οργανώθηκε από το ανώτατο στρατηγείο του Νόρφολκ και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Στρατηγείου του Στεφάν Αμπριέλ έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική μας και να ελέγξουμε καλύτερα τους στόχους μας σε σχέση με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Καζακστάν, της Αυστραλίας και εταίροι δηλαδή της συμμαχίας, όχι μόνο μέλη. Όσα τα Ηνωμένα Έθνη, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και εκπρόσωποι του τύπου, σημαντικοί εκπρόσωποι του τύπου. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων συναντήθηκε και με πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μέλη πολλών κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι δικές σας απόψεις ε, ε, ελήφθησαν υπόψη. Ένας άλλος πολύ σημαντικός στόχος είναι να γίνουν γνωστές αυτές οι προσπάθειες. Η στρατηγική αντίληψη, έλεγαν οι Αμερικανοί, θα πρέπει να είναι αναγνώσιμη σε όλο τον κόσμο και στον κοινό άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και στον Πολωνό υδραυλικό. Νομίζω ότι έτσι θα φέρουμε τα στοιχεία αυτής της συζήτησης και σε ένα ευρύτερο κοινό. Ξεκινήσαμε με 12 εμπειρογνώμονε, καταλήξαμε με 10 γιατί ο ένα πήρε προαγωγή και ασχολήθηκε με άλλα θέματα. Ε, καταλήξαμε σε ένα πολύ συνοπτικό κείμενο 64 σελίδων και τώρα έχουμε άλλη μία προσπάθεια το πώς να περάσουμε από την έκθεση αυτή της στρατηγικής ε, στη συγκεκριμένη έννοια. Κατά κάποιο τρόπο βρισκόμαστε σε μία δεύτερη φάση θα έλεγα όπου ο Γενικός Γραμματέας προσωπικά θα προετοιμάσει ακριβώς το έγγραφο αυτό. Και επίσης οι συνάδελφοι από το Διεθνές Προσωπικό της Συμμαχίας θα τον υποστηρίξουν. Ο Γενικός Γραμματέας θα δημοσιεύσει το κείμενο αυτό πριν από το τέλος του Σεπτεμβρίου. Θα γίνει μια πρώτη κοινή συζήτηση Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας τον μήνα Οκτώβριο στις 14 του μηνός είναι το λεγόμενο Τζάμπο Συμβούλιο και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα υιοθετήσουν το τελικό κείμενο στη Λισαβόνα τον Νοέμβριο, στις 19 Νοεμβρίου. Τώρα τι μορφή θα πάρει το τελικό κείμενο αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 10 σελίδες, θα είναι ένα πολύ ανοιχτό και δεκτικό κείμενο και μετά από την αντίληψη αυτή την κοινή της στρατηγικής στην οποία καταλήξαμε, ρόλος μας και ρόλος των στρατιωτικών συμβούλων είναι να ε, προσφέρουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση η οποία θα μας οδηγήσει ε, στο να αποκτήσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα που θα μετατρέψει αυτή την γενική γλώσσα σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα καθοδηγήσουν τη δράση μας στο μέλλον. Θα ασχοληθούμε με τα θέματα των ικανοτήτων της Συμμαχίας των Στρατιωτικών, κάποια προγράμματα τα οποία πρέπει να υιοθετήσουμε ή όχι κτλ. Και φυσικά εδώ η σημασία των σχέσεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτεύουσα και η Προεδρία μας τον επόμενο χρόνο θα έχει το θέμα αυτό σαν μια βασική προτεραιότητα. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη, την κυρία Ανδρεανή τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω στην παρουσίαση που έκανε ο Πολωνός πρέσβης. Έχει ανοίξει πια η διαδικασία. Όπως είπε βρισκόμαστε σε μια δεύτερη φάση τώρα, περιμένοντας από το Γενικό Γραμματέα να μας παρουσιάσει το κεντρικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι η βάση του εγγράφου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Λισαβόνα. Να υπογραμμίσω ποια είναι για μας και ομιλώ εξ ονόματος της Γαλλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι τα σημαντικά θέματα για τη Λισαβόνα. Πρώτον, πιστεύουμε να υπάρξει μια συμφωνία. Στο ΝΑΤΟ όλα πηγαίνουν με συνένεση και πρέπει να υπάρξει μια συνένεση. Αυτή η συνένεση σήμερα δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά λοιπόν. Δεύτερον, κάτι το οποίο συνδέεται με την έννοια της στρατηγικής αντίληψης και όχι μόνο. Ελπίζουμε χάρη σε αυτή τη στρατηγική αντίληψη να ξεκινήσει μια πραγματική διαδικασία μεταρρύθμισης. Υπάρχει το οικονομικό πλαίσιο το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Θέλουμε να καταστήσουμε πιο ορθολογική την εργασία μας, να μεταρρυθμίσουμε και την έδρα και το στρατηγείο και θα πρέπει ακριβώς αυτή η στρατηγική αντίληψη να μας βοηθήσει να το πετύχουμε. Τρίτον, στα πλαίσια των θεμάτων τα οποία συζητάμε, Θέλουμε, χάρη πάντα σε αυτήν τη συνένεση, να καταλήξουμε σε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στο άρθρο 5 της Συμμαχίας της συλλογική Άμυνας και τη διαχείριση των κρίσεων. Σήμερα το ΝΑΤΟ ξέρετε ότι είναι στο Αφγανιστάν και θα πρέπει να βρεθεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά. Για τη Γαλλία ένα βασικό θέμα λοιπόν της συλλογική άμυνας είναι η αποτρεπτική ικανότητα της συμμαχίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο τελικό έγγραφο. Τελευταίο σημείο, οι εταιρικέ σχέσεις. Επιμένουμε σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις. Είναι ένα επιπλέον νέο στοιχείο, στο οποίο θεωρούμε ότι έχουμε συμφέρον να προχωρήσουμε. Η προηγούμενη συμφωνία έχει ηλικία άνω των 10 ετών. Υπάρχει η Ρωσία, βασικό θα έλεγα συστατικό, οι υπόλοιποι εταίροι μας, όπως τους ονομάτισες κάποιους από αυτούς, και οι υπόλοιπε διεθνείς οργανώσεις και ε, ε, επικεφαλής όλων αυτών των διεθνών οργανώσεων φυσικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέση ΝΑΤΟ ευρωπαϊκή ένωση Ο Γενικός Γραμματέας Σάσμουσεν εξεφράστη στην αρχή της εβδομάδας γύρω από το θέμα αυτό. Ήδη από τη στιγμή που ανέλαβε είπε ότι είναι βασική προτεραιότητα αυτή Έχουμε εμπλακεί στα ίδια θέατρα επιχειρήσεων, Κωσυφοπέδιο, Αφγανιστάν, καταπολέμηση της πειρατείας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη σχέση αυτή ακόμα περισσότερο. Για τη Γαλλία αυτό θα είναι το βασικό αποτέλεσμα το οποίο περιμένουμε να πετύχουμε. Ελπίζω οι ερωτήσεις να δώσουν λαβή σε ε, συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Άρχισα να φοβάμαι λίγο όταν είδα τον Τζέφρι Βαν Όρντεν να βάζει ακουστικά με το που άρχισα να μιλάω στα αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, τις ευχαριστίες μου, αλλά και την ανησυχία μου επειδή με προσκαλείτε για δεύτερη φορά εδώ. είτε επειδή ήμουνα τόσο πιστικό την πρώτη φορά και την δεύτερη φορά περιμένετε μία πολύ καλή επανάληψη της προηγούμενης παράστασης, είτε ήμουνα πάρα πολύ κακό την πρώτη φορά και περιμένετε τώρα μπας και καταλάβετε κάτι περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, θα σας ενημερώσω σήμερα για το τι κάνει το άλλο θεσμικό όργανο που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στο ΝΑΤΟ. Καταρχάς, να σας μιλήσω για τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη στρατηγική μας. Τρία βασικά πράγματα. Όταν προσπαθείτε να κάνετε μία μεταρρύθμιση ενός οργανισμού. Τότε δεν μιλάμε απλά για ένα χαρτί, αλλά για μια διαδικασία. Και γι' αυτό πρέπει να μπορούμε να απομακρυνθούμε από τα καθημερινά και να εξετάσουμε τι θα έπρεπε να κάνουμε, έτσι ώστε να ισχύουν αυτά και μετά από 5 ή 10 χρόνια. Οπότε προκύπτουν τα εξής ερωτήματα. Καταρχάς, τι δεν κάνουμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να κάνουμε. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Δεύτερο ερώτημα. Τι άλλα πράγματα επιπλέον πρέπει να κάνουμε για να παραμείνουμε ζωτικοί για τον 21ο αιώνα. Και τέλος, τι διάρθρωση, τι διαρθρωτική δομή χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα σύστημα που θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Πολλοί οργανισμοί, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζουν χάσμα μεταξύ των φιλοδιοξιών τους και των πόρων τους. Βεβαίως, ε, οι οργανισμοί ασφαλείας ίσως δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Τώρα, όπως γνωρίζουν και οι Σοφοί και η Επιτροπή υπό την ηγεσία της κυρίας Όλμπραϊτ, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουμε εντοπίσει ως βασικά. Καταρχάς, το άρθρο 5. Τι σημαίνει με την παραδοσιακή έννοια ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις στο έδαφος μας είναι μια πραγματική δέσμευση η οποία βασίζεται στην ετοιμότητα των δυνάμεων, στον ασκήσεις που γίνονται κτλ. κτλ. Όμως, μέσω των αλλαγών που έγιναν το 2001, μπορεί το άρθρο 5 να χρησιμοποιηθεί και για μη παραδοσιακά σενάρια, για μη παραδοσιακές επιθέσεις. Για παράδειγμα, τρομοκρατικές επιθέσεις ε, κυβερνοεπιθέσεις, ε, όλα αυτά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο άρθρο 5. Βεβαίως αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των συμμάχων, αλλά δεν μπορούν να αποκλειστούν αυτά τα ενδεχόμενα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αυτά. Δεύτερον, τι σημαίνει ο όρος αποτροπή για τον 21ο αιώνα και τις προκλήσεις του κάποια πράγματα που λειτουργούσαν επιτυχώς στο παρελθόν μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά και στο μέλλον. Και το ΝΑΤΟ διαθέτει ένα μείγμα συμβατικών και πυρηνικών δυνάμεων, αλλά το ερώτημα είναι αν χρειαζόμαστε και άλλες δυνατότητες αποτροπής. Για παράδειγμα, μέσω μιας καλύτερης διαχείρισης κρίσεων και καλύτερης πρόληψης συγκρούσεων. Μιλάμε δηλαδή για στοιχεία που δεν θα αντικαταστήσουν το μείγμα πυρηνικών και συμβατικών μέσων που διαθέτουμε, αλλά θα τα συμπληρώνει. Επίσης, το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι είναι και φορέας διαβούλευσης διατλαντικής. Όμως, Υπάρχει η εντύπωση ότι πλέον ασχολούμαστε περισσότερο με επιχειρήσεις και ότι οι διαβουλεύσεις συνήθως γίνονται μετά την έλευση του στρατού και όχι πριν. Αυτό έγινε στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα. Υπήρχαν και επιχειρήσεις ε, στα Βαλκάνια και στο κόλπο του Άντεν. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε μία πιο ευρία αντίληψη πλέον και επομένως έναν πιο ευρύ ορίζοντα για τις διαθλαντικές επιχειρήσεις. Η έκθεση Albright μιλάει για μεγαλύτερη χρήση του άρθρου 4, προτείνει μεγαλύτερη χρήση του άρθρου 4. Κάτι που θα μπορούσε, αλλά ίσως και όχι να είναι η κατάλληλη οδός. Ίσως όμως δεν θα έπρεπε να επικεντρωνόμαστε στα άρθρα. Το βασικό είναι να χρησιμοποιήσουμε το ΝΑΤΟ περισσότερο ως διακλατικό φόρουμ. Να υπάρχει μία ανοιχτή πόρτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε μια έντονη διεύρυνση τα τελευταία χρόνια που ενδεχομένως να μην συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς στο μέλλον για τους γνωστούς λόγους, όμως, ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τονίσουμε ότι οι πόρτες του ΝΑΤΟ παραμένουν ανοιχτές σε όλους τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια. Και περνάω πάλι στο ερώτημα του τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα, που ανέφεραν και οι πρέσβεις. Προφανώς, η στρατιωτική πτυχή είναι βασικό κομμάτι, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Διαπιστώσαμε στο Αφγανιστάν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικές από ό,τι θα έπρεπε όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πώς λοιπόν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα λειτουργεί καλύτερα για το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να έχουμε κάτι το ολοκληρωμένο από την αρχή και όχι μόνο αφού σε ε, κατέβουν τα στρατεύματα. Και αυτό θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια μιας καλύτερης συνεργασίας και στοιχείων που θα μπορούσαμε να μας βοηθήσουν να συνεργαστούμε περισσότερο ενδεχομένως θα έπρεπε να αποκτήσει ορισμένες πολιτικές δυνατότητες, πολιτικά μέσα το ΝΑΤΟ, όχι για να υποκαταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να μπορεί να συμπληρώσει άλλους οργανισμούς ή ενδεχομένως για να μπορεί να καλύπτει ένα προσωρινό κενό που μπορεί να υπάρχει μέχρι να έρθουν άλλες πολιτικές οργανώσεις, άλλοι πολιτικοί οργανισμοί. Και τι θα πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο, τι πρέπει να αυξήσουμε. Ένα βασικό θέμα εδώ είναι οι προκλήσεις ασφαλείας που υπάρχουν σήμερα. Για παράδειγμα, κυβερνοεπιθέσεις, τρομοκρατία, θέματα ενεργειακής ασφάλειας, πυρηνικών όπλων, πρόκειται για πραγματικές προκλήσεις για τους συμμάχους μου. Από την άλλη, στιγμή, από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι πρώτον δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα και δεύτερον χρειαζόμαστε πολύ καλούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν είναι αποκλειστικά στρατιωτικοί. Το ΝΑΤΟ θα είναι επιτυχές μόνο αν έχει τις κατάλληλε εταιρικές σχέσεις για παράδειγμα. Αν έχουμε κάποια στιγμή μια κύβερνο επίθεση, πρέπει να έχουμε τα μέσα για να ανταποκριθούμε. Και δεύτερον, κάτι που ανέφερε επίσης ο πρέσβης Αντριάνη, αφορά το θέμα της πρόληψης. Λυπάμαι που το λέω, αλλά κάποιες από τις πιο χρεωμένες χώρες στον κόσμο που υποφέρουν περισσότερο από την οικονομική κρίση είναι οι εταίροι μας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Άρα, ίσως θα έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν είχαμε προβλέψει αυτή την κρίση και ίσως θα χρειαστούμε δισεκατομμύρια για να την αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτό τι μας διδάσκει ότι η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη. Τέλος. Στη λειτουργία μας εντός της Ευρώπης και στην αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν όλο τον κόσμο και όχι μόνο τον ΝΑΤΟ, όπως παλιά ο ψυχρός πόλεμος, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τους εταίρους μας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τι θα κάνουν αυτοί για εμάς, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς. Τέλος, επειδή ήδη αναφέρθηκε, δεν αξίζει τον κόπο να έχουμε έναν οργανισμό του 20ου αιώνα για τις προκλήσεις του 21ου. Και εγώ που ασχολούμαι με τον ΝΑΤΟ από το 1980, θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές, αλλά και πολλά πράγματα που εξακολουθώ να τα αναγνωρίζω. Αν είχα μπει σε μία μηχανή του χρόνου το 1980 και είχα έρθει στο 2010, θα αναγνώριζα πολλά πράγματα σήμερα από το παρελθόν. Άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πολλά από αυτά τα πράγματα για τη μεταρρύθμισή μας. Σήμερα το πρωί είχαμε μία συνάντηση με τους πρέσβεις για ένα πολύ βασικό θέμα, την, ε, τον καλύτερο συντονισμό πληροφοριών του ΝΑΤΟ έτσι ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε καλύτερα την κατάσταση επιτόπου πριν εμπλακούμε. Επίσης, πρέπει το προσωπικό να ασχολείται περισσότερο με τις προτεραιότητες. Γιατί αυτή τη στιγμή ίσως να έχουμε περισσότερο άτομα στο προσωπικό να ασχολούνται με χαμηλού επίπεδου προτεραιότητες. Τώρα άλλα θέματα κοινή χρηματοδότηση, για παράδειγμα, των επιχειρήσεων. Αν πρέπει να έχουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εκτός των συνόρων μας, τότε χρειαζόμαστε και μία κατάλληλη οργανωτική δομή και θα πρέπει το ΝΑΤΟ να είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτή θα είναι μια βασική πρόκληση για το ΝΑΤΟ μετά το Αφγανιστάν. Πρέπει μεν να γίνουν περικοπές, αλλά με τον κατάλληλο τρόπο και να διαχειριστούμε τις ε, μειώσεις των προϋπολογισμό με τρόπο που θα εξακολουθεί να επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν και το ΝΑΤΟ να συμμετέχει σε αυτές τις συζητήσεις και όχι απλά να παρατηρεί τις εξελίξεις της πρωτεύουσα. Αν κάνουμε προσεκτικά κάποια βήματα, χωρίς να υπερφορτώσουμε το ΝΑΤΟ και αν βρούμε την κατάλληλη δομή, τότε θεωρώ ότι η νέα στρατηγική δεν θα είναι απλά ένα κομμάτι χαρτί. Ευχαριστώ. Να σας διαβεβαιώσω ότι ο λόγος που σας προσκαλέσαμε ξανά είναι γιατί πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας. Ζαν Φρασουά, παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία. Ο Τζέιμι μίλησε για το πλαίσιο. Εγώ καταρχάς να επιμείνω σε κάτι σημαντικό που ζητούσαμε από την αρχή. στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Μία δημόσια συζήτηση για το θέμα. Διαφάνεια. Ε, κατά την εξέλιξη των συζητήσεων αυτό είχε συγκεκριμένες συνέπειες. Συμφώνησαν ε, ο Γενικός Γραμματέας, η κυρία Όλμπραϊτ και η ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα τέλη Αυγούστου ότι θα υπήρχε μία συζήτηση επί της βάσης όπου θα προσπαθούσαμε να θέσουμε τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο των σημερινών απειλών. Και αυτό που υπονοείται εδώ είναι ότι τα θέματα της ασφάλειας, τρομοκρατία, άμυνα κτλ. θα πρέπει να τα δούμε και να τα πούμε στους πολίτες. Γιατί οι πολίτες ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα και ως φορολογούμενοι, αλλά και επειδή τους αφορούν τους ίδιους πραγματικά, αν και ενδεχομένω δεν αφορούν την απλή καθημερινή τους ζωή. Το 99 στο προηγούμενο στρατηγικό συμβούλιο υπήρχε ο στόχος η συζήτηση να φτάσει σε όλους τους πολίτες. Τώρα, δεν θα μιλήσω βεβαίως α, λεπτομερές για τα έγγραφα. Θα πω όμως ότι αυτά δημιουργήθηκαν μετά από μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαν ε, φοιτητές, ε, κυβερνήσεις, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι οποίοι όλοι ασχολήθηκαν με τα θέματα της στρατηγικής. Είχαμε λοιπόν πολίτες που συμμετείχαν στη συζήτηση, την κοινωνία των παλιτών. Τώρα, η πρώτη εκτίμηση για αυτή τη συζήτηση. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Πρέπει να βελτιώσουμε και να τονίσουμε τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, συνειδητοποιούμε ότι ειδικά οι νέοι ανησυχούν για τις συνέπειες της αυξημένης πολυπλοκότητας της άμυνας και της ασφάλειας. Είτε μιλάμε για τρομοκρατία, είτε για κυβερνοασφάλεια. Τα θέματα αυτά δεν τους φαίνονται πλέον απλά και πρέπει να υπάρξει διαπαιδαγώγηση για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά. Εμείς θεωρούμε ότι η έγκριση τη στρατηγικής από τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα είναι απλά ένα βήμα στη διαδικασία προκειμένου στο επόμενο βήμα να περάσουμε στους πολίτες και την κοινωνία. Δεύτερο θέμα, κοινή γνώμη. είναι προφανές ότι η άμυνα και η ασφάλεια δεν θεωρούνται και για την κοινή γνώμη. Όλοι γνωρίζουν τις απειλές και από τους διάφορους μηχανισμούς μας διαπιστώνουμε ότι για πολλούς εταίρους μας στη συμμαχία υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια. Αν και βεβαίως αυτή η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πάντως, μεταξύ των ερωτημάτων που πάντα τίθενται, ένα από τα βασικότερα είναι το πώς μπορεί να υπάρξει η καλύτερη συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το θέμα που κυριαρχεί συνήθως για τους πολίτες και το οποίο δεν γίνεται κατανοητό στους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν υπάρχουν πιο απτές αποδείξεις αυτής της συνεργασίας. Ένα δεύτερο θέμα αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία. Μπορεί να γίνει μια αναπαράσταση της ε, ασφάλειας ολόκληρης της Υπήρου και εκεί οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι ένα βασικό θέμα για το οποίο τίθενται συνεχώς ερωτήσεις. Οι σχέσεις λοιπόν με τη Ρωσία και οι απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στο πλαίσιο της στρατηγικής θα έχουν συνέπειες για το μέλλον της συμμαχίας μετά. Έρχονται οι σχέσεις του ΝΑΤΟ με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ο Τζέιμι μας υπενθύμησε ότι το ΝΑΤΟ δεν θέλει να γίνει ο παγκόσμιος χωροφύλακας. Όμως πρέπει να δούμε τι σχέσεις θα έχουμε με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, στενές ή όχι, αλλά με πολλούς οργανισμούς όπως το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα θέματα που τίθεται συχνά. Αυτό το θέμα απασχόλησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Θεωρούμε ότι και εκεί πρέπει να υπάρξει διαπαιδαγώγηση του κοινού και κάτι που θα έπρεπε να επιδιώξουμε περισσότερο είναι να εξετάσουμε και την στρατηγική ασφαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για το μέλλον. Τι ομοιότητες ή παραλληλισμοί μπορούν να υπάρξουν. Η ευρωπαϊκή ιδέα για την ασφάλεια όπως μεταρρυθμίστηκε το 2008, θεωρούμε ότι έχει συνέπειες και για εμάς. Είπα και πριν ότι ο Γενικός Γραμματέας θέλει να καταλήξει σε ένα έγγραφο σύντομο και σαφές. Έτσι ώστε να μπορούμε να περάσουμε ένα κεντρικό μήνυμα προς όλους ότι η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι κεκτημένα, ότι εξακολουθούν να απαιτούνται προσπάθειες για την άμυνα και την ασφάλεια και υπενθυμίζω ότι εξαιτία της οικονομικής κρίσης μπορεί να έχουμε δυσκολίες στο να δείξουμε τη χρησιμότητα μιας ε, συνεχιζόμενης αμυντικής προσπάθειας και στο μέλλον. Ίσως θα ήταν δύσκολο να περάσουμε αυτό το μήνυμα, αλλά εγώ παρόλα αυτά θα ήθελα να το περάσω σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον ε, Ντάριος Βόλκισκη, πρόεδρο της αντιπροσωπείας για τον ΝΑΤΟ. C'est une Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν μια αντιπροσωπεία με έναν ε, εταίρο καθόλου εύκολο. Εγώ έχω αναλάβει την Προεδρία της Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ και ήμουν στη Ρίγα και έπρεπε να αναρωτηθώ σαν το Σέξπιρ να ζει κανείς ή να μην ζει. Είναι πολύ δύσκολη λοιπόν η δουλειά. Αλλά να περάσω κατευθείαν στο ερώτημα τι μπορεί να φέρει, τι καινούργιο μπορεί να φέρει η σχέση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μπορεί να έχει κάποια προστιθέμενη αξία, γιατί προς το παρόν αυτά τα πράγματα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ό,τι και αν αναφέρεται στο κείμενο του Σολμπράιτ. Δείχνει ότι Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει το ΝΑΤΟ των Βρυξελών και υπάρχει η Ευρώπη, τον Ευρωπαϊκή Ένωση των Βρυξελών. Και δεν θυμάμαι ποτέ καμία συνάντηση με βασικούς, σε επίπεδο ας πούμε βασικών εξαρχουσών προσωπικότητων από αυτή, ε, σε τέτοιο επίπεδο ε, από τους δύο αυτούς οργανισμούς. Έχουμε και την έκθεση Βάτανεν Βέβαια, πολλέ φορέ μόνο οι Γάλλοι μπορούν να είναι τόσο ευρηματικοί. Ε, είναι αυτό που σα κάνω, δεν το λέω. Μην με παρεξηγήσετε. Όλο συζητούμε, όλο. Και ο Σολάνα επίση ήταν γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και τώρα είναι ο ύπατος εκπρόσωπο. Ε, πρέπει να λέμε λίγο τα πράγματα και με το όνομά τους πριν ξεκινήσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον. Uh, Εγώ διάβασα το κείμενο. Εντάξει, για δημόσιες σχέσεις είναι καλό, αλλά μέσα στις δέκα σελίδες πόσες γραμμές υπάρχουν αφιερωμένες στις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το δυο, τρεις, τρεις. Τα πάντα έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία και με την πολιτική βούληση. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές οπτικές, δύο διαφορετικά πολιτικά οράματα και φιλοσοφίες. Και δεν είναι και κατά τύχη και συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στην Επιτροπή του, που έχει προσκαλέσει Γάλλους και Πολωνούς ε, ε, ε, πρέσβεις. Είναι τα μόνα κρατημέλη που τονίζουν την αναγκαιότητα της σύγκλησης απόψεων και της συνεργασίας για θέματα ασφάλειας. Ούτως ή άλλως αυτό είναι και από τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Πολιτική βούληση λοιπόν και φιλοσοφία. Και επίσης θα έπρεπε να ζητήσουμε να υπάρξει αυτή η δράση. Ούτω ή άλλω όλοι οι ίδιοι πολίτε είμαστε. Είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέλη και στην ΝΑΤΟ μέλη. Πριν από δύο χρόνια νομίζω είχαμε κάνει, είχαμε αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρημα. Δύο χρόνια νομίζω. δεν έφταιγε το ΝΑΤΟ που ζήτησε την στενότερη ε, συνεργασία, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχα πάει στα κεντρικά της, ε, του ΝΑΤΟ στον ε, Γιάνν Χούμπ Σέφερ με τον Πέτεριν και τον Φον Βόγκαου και τους εκπροσώπους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και είχαμε πει να καλέσουμε τον Γιάνν Χούμπ Σέφερ να έρθει και δεν ήρθε ποτέ. Ποτέ δεν ήρθε. Τώρα περιμένουμε τον Ράσμουσεν. και με την δική μου ε, πρωτοβουλία η ΑΦΕΤ ε, και η Επιτροπή Άμυνας ε, τον έχει προσκαλέσει. Τώρα θα έρθει να έρθει να δει τον Μπούζετ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια κοινή τέτοια συνεδρίαση για, μεταξύ αυτών των επιτροπών για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Οπότε αν μπορείτε ε, του την επιθυμία μας το Φλεβάριο του 2009 όταν ήμουν πρόεδρο, συζητήσαμε το θέμα αυτό και βελτιώσαμε την πρώτη έκθεση Βάτανεν. Θα θυμάστε κυρία Γκόμε. Και μετά πήγα στο Δημβούργο. Και ζήτησα, ε, μάλιστα, μάλλον μίλησα με πολλού ε, από τον ΝΑΤΟ, στρατιωτικού και μη. Κανένας δεν είχε ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ή ε, τέλο πάντων εντάξει, μπορεί να το έχει ακούσει, αλλά το, η έκθεση του Κοινοβουλίου για, την, για τι σχέσει ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση τίποτα δεν είχαν ακούσει. Ακόμη και αυτοί που έγραφαν τι δηλώσει κτλ. Τίποτα δεν ήξεραν. Και ξανακοίταξα, το ξαναρώτησα και στη Ρήγα. Το ίδιο πράγμα. Κανεί δεν ήξερε. Ούτε κανένα είχε διαβάσει την έκθεση. Ούτε ήξερε ότι υπάρχει έκθεση τέτοια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν δηλαδή κάτι που δεν το κατάλαβε καν το ΝΑΤΟ. Otherwise I wouldn't even know that you are here. Ευτυχώς δηλαδή σήμερα που είχαμε αυτή την κοινή συνεδρίαση, γιατί αλλιώς ούτε καν θα ήξερα ότι είσαστε εδώ. Χρειαζόμαστε πιο στενές σχέσεις, όχι ανταγωνιστικές. Οι εμπειρογνώμονες μπορούν να μας πούνε πώς θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και προς τον παρόν δεν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Δεν θέλω βέβαια να είμαι μόνο επικριτικός, αλλά πρέπει να πω και κάποια καλά λόγια για το ΝΑΤΟ. Πρώτη φορά το ΝΑΤΟ ήταν ο οδηγός μας όταν ε, εκπονήσαμε το ψήφισμα το καλοκαίρι του 2009 για τη Γεωργία που ακολούθησε τις θέσεις του ΝΑΤΟ. Πρώτη φορά λοιπόν ε, συμφωνούμε απόλυτα με την ε, θέση του ΝΑΤΟ στην, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Εν συντομία θα έλεγα ότι ακούμε αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να αλλάξουμε και θα ήθελα να δούμε και τα θέματα συνεργειών, να δούμε πώς μπορούμε να γκρεμίσουμε τα τείχη μεταξύ αυτών των δύο οργάνων και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, συνεργασία μεταξύ μας. Όλα αυτά πρέπει να οριστούν σαφέστερα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι το νέο στρατηγικό συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι υπάρχει πτυχή ασφαλείας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας που στόχος της είναι να βελτιώσει και τις υποδομές ασφαλείας και τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπληρώσει τις συνατοικές δυνάμεις. Όλα λοιπόν είναι μπροστά μας ακόμα. Ελπίζω να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Προς το παρόν είπαμε πώς έχει η κατάσταση και για τις δύο πλευρές. Ε, μάλλον τώρα θα αρχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Ναι, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνέργεια, συνεργασία ε, και δεν γίνεται τίποτα τελικά. Μόνο τα λέμε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Και δεν θα έπρεπε. Όταν ε, ήμασταν στο Εδιμβούργο, είπαμε, εσείς συνάδελφοι από το ΝΑΤΟ, περιμένετε κάτι από μας μια συμβολή, δεν μας έδωσε κανένας καμία απάντηση. Μόνο έκπληξη είδαμε στα πρόσωπα όλων. Ήμασταν, πώς μας λένε, συνδεδεμένοι, πώς μας λένε, τι καθεστώς έχουμε μαζί με τους Παλαιστινίους, τους Ιρανούς. Ναι, στο η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ίδιο καθεστώς με το Ιράν. Δεν θα ε, ξεκινήσετε πόλεμο με το Ιράν, έτσι. Τούτη τη βδομάδα τουλάχιστον όχι. Οπότε το θέμα είναι πώς μέσω αυτή της νέας ε, στρατηγικής και της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας θα ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Έτσι δεν είναι. Από την πλευρά της Ένωσης Φυσικά πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αυτού του άρθρου 5 και του κλασικού ρόλου που έχει να παίξει το ΝΑΤΟ και των νέων προκλήσεων που υπάρχουν εκτός της Ευρωατλαντικής του ευρωατλαντικού χώρου. Φυσικά μας ενδιαφέρουν οι μη συμβατές, ε, συμβατικές ε, επιθέσεις, όπως ας πούμε μια επίθεση στο διαδίκτυο στο ΝΑΤΟ μας είπανε ναι ωραία εντάξει να γίνει η έκθεση και εμεί είπαμε στην εξωτερικών υποθέσεων να κάνουμε την έκθεση και δεν έγινε ποτέ η έκθεση. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε τα έγγραφα που ζητούμε, είπαμε εμεί στο ΝΑΤΟ, τίποτα δεν μας έστειλαν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον. Ε, ε υπήρχαν οι υποσχέσεις, αλλά δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα τελικά νέες προκλήσεις. Ε, πειρατεία από τη Σομαλία, κυβερνοπειρατεία, ε, όλα αυτά πρέπει να απαιτούν να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες. Πρέπει να συνεργαστούμε. Γιατί αυτό που κάνουμε τώρα καλό είναι, αλλά δεν είναι αρκετό. Τα νέες προσδοκίες της Ένωσης τις ξέρετε. Για να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. να δούμε τι θα γίνει και με το γαλλοπολωνικό όραμα. Έχουμε όμως, νομίζω, να συμβάλλουμε, έχουμε μεγάλο ρόλο να παίξουμε, να βοηθήσουμε τον ΝΑΤΟ. Διορθώνοντας λίγο αυτή την ε, αίσθηση ανικανότητας που υπήρχε με το Αφγανιστάν, για πολύ σημαντικά θέματα, όπως κάτι που έχει συζητηθεί και στην Επιτροπή Πολιτισμού εδώ, με πρόεδρο την Doris Πακ για τις ε, διανέξεις και το πώς μπορούν να λυθούν. Το έχετε σκεφτεί αυτό εσείς ποτέ στο ΝΑΤΟ. Και συνεχίζω στα γαλλικά. Η νατοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για και αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, δεν ξέρω. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ευρω... εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αλλαγή πνευματική, φιλοσοφική. Διαφορετικά οι επαναλήψεις δεν μας οδηγούν πουθενά. Άρα Αναμένουμε με ενδιαφέρον την επίσκεψη Ράσμουσεν. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ευγένεια, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε. Το ελάχιστο είναι ότι θα υπάρξει συζήτηση για την αμοιβαία μας σχέση εδώ στο Κοινοβούλιο. Και μετά την συνθήκη της Λισαβόνας, ίσως κάτι τέτοιο θα ήταν λογικό. Βεβαίως ε, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τις ε, στρατηγικές πριν τη Λισαβόνα, τη δική σας Λισαβόνα, πριν οριστικοποιηθούν όλα εκεί. Άρα, ας κάνουμε κάτι και σύντομα. Διαφορετικά, σε ένα χρόνο θα ξαναβρισκόμαστε για να λέμε τα ίδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους κυρίους πρέσβεις, τον Τζέιμι Οσέι και τους πρέσβεις επαναλαμβάνω για την παρουσία τους εδώ και για τη διαθεσιμότητά τους να συζητήσουν τις νέες στρατηγικές αντιλήψεις για τον ΝΑΤΟ και να συνεχίσουμε μια συζήτηση την οποία είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε στο παρελθόν με την κυρία Όλμπραϊτ και τώρα οι συζητήσεις δράζονται σε ένα συγκεκριμένο κείμενο. Νομίζω ότι το κείμενο αυτό είναι ισορροπημένο κείμενο, ίσως πολύ ισορροπημένο, γιατί ε, κρατάει ανοιχτές περικές φορές πολλές επιλογές, κάτι το οποίο ίσως σε αυτή την προκαταρκτική φάση είναι απαραίτητο ή αναπόφευκτο. Υπάρχουν όμως θετικά βήματα σε σχέση με το στόχο μας, που δεν είναι να επανεφεύρουμε τον ΝΑΤΟ, αλλά να ανακαλύψουμε τον ΝΑΤΟ. Να ανακαλύψουμε τον ΝΑΤΟ μετά από προβληματικά χρόνια που εξασθένησαν την συμμαχία και εξασθένησαν επίσης και τον διατλαντικό θεσμό γενικότερα. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και ορισμένες ερωτήσεις να θέσω. Πρώτον, σχετικά με τις πολιτικές ικανότητες ή καλύτερα τις μη μάχινες, μη στρατιωτικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Εφόσον πάντα παραμένουν ε, ε, ορατές συγκεκριμένες απειλές και απαραίτητες ορισμένες απαντήσεις, ε, ανταποκρίσεις θα έλεγα σε αυτές τις απειλές. Η έννοια της συμπληρωματικότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ΚΕΠΑ Εν πολλής μου φαίνεται ότι αμφισβητείται από τις προσπάθειες τις οποίες κάνει το ΝΑΤΟ σε επίπεδο μη ε, στρατιωτικών παρεμβάσεων. Έχουμε να κάνουμε με ένα ΝΑΤΟ το οποίο θέλει να ασχοληθεί και με τη μη στρατιωτική διάσταση. Θέλουμε ένα ΝΑΤΟ το οποίο να ασχολείται όλο και περισσότερο με ένα πρόβλημα το οποίο είναι όλο και πιο σημαντικό. Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα της αποτροπής. Το θέμα της αποτροπής, ίσως μάλλον ο τομέας της αποτροπής στο έγγραφο αυτό, ίσως να μην είναι ο πιο ισορροπημένος από τους υπόλοιπους τομείς τουλάχιστον, ε, όταν συζητιέται ένα θέμα όπως ο ρόλος ε, της ε, μη στρατηγικής πυρηνικής δύναμης, της τακτικής στρατιωτικής, ε, μάλλον πυρηνικής δύναμης, ακούγονται κάποια επιχειρήματα τα οποία δεν είναι θα έλεγα ιδιαίτερα υποστηρίξιμα σχετικά με την χρησιμότητα ύπαρξης αυτού του είδους της αποτροπής και λόγω του πολιτικού ρόλου τον οποίο τελικά έχουν αυτά τα όπλα μου φαίνεται ότι η τεκμηρίωση η οποία υπάρχει δεν είναι επαρκής. Τέτοιου είδους όπλα γεννιόνται θα έλεγα με αυστηρά πολιτικά κριτήρια, θυμόμαστε τον Κίσιντζερ είναι κάτι το οποίο μπορεί να απελευθερώσει αν θέλετε ένα μεγαλύτερο πεδίο δράσης για την διπλωματία και την εξωτερική πολιτική εφόσον δεν τίθεται θέμα μαζικής στρατιωτικής απάντησης, ανταπόδοσης αλλά παρόλα αυτά το θέμα της τακτικής πυρηνικής δύναμης είναι κάτι το οποίο ανεπαρκώς τεκμηριώνεται στο έγγραφο αυτό που όπως ε, είπαμε είναι κάτι το οποίο ε, μερικές φορές θα πρέπει να τεθεί σε συζήτηση όχι μόνο στις χώρες οι οποίες είναι πυρηνικές δυνάμεις αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, στις γειτονικές χώρες. Εγώ ήμουνα φυσικά παρατηρητής στη Ρήγα ενώ αντίθετα ο Ζιρινόφσκι σαν παράδειγμα ήταν πλήρες μέρους της ε, συζήτησης, του σώματος το οποίο οργάνωσε τη συζήτηση. Έχετε ακούσει και τα της εκθέσεως Νόξου, ξέρετε ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με αρκετά καλό τρόπο, έτσι ώστε να διευκρινιστεί η πολιτική του ΝΑΤΟ σε τομείς, ε, επαναλαμβάνω, όπως τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Νομίζω ότι ένα βασικό θέμα σχετικά με την πυραυλική άμυνα, μια διάσταση την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, είναι να διαπιστώσουμε ότι πέραν των τεχνικών προβλημάτων τα οποία παραμένουν χαίνοντα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα πολιτικά τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα και θα πρέπει να μας καταστήσουν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν υπάρξει νέα χαρακτηριστικά στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική, ακόμα και την κοινή εξωτερική πολιτική. Και νομίζω ότι έχει αρκετά μεγάλη σημασία η αλλαγή αυτή και αυτό δεν φαίνεται εύκολα στο κείμενο. Και η παράγραφος αυτή δεν παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο συγκεκριμένο έγγραφο και δεν θα έλεγα τεκμηριώνει με σωστό τρόπο το θέμα της συμπληρωματικότητας η οποία θα πρέπει να συζητηθεί σε βάθος και εφόσον πράγματι θέλουμε να μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτής της νέας στρατηγικής αντίληψης το θέμα αυτό θα συζητηθεί πολύ περισσότερο ακόμα και σχετικά με την αναγνώριση της σημασίας που έχουν ε, οι ρόλοι πολιτικοί και στρατιωτικοί που μπορεί να αναλάβει η Ευρώπη. Κύριος Βανόρντεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη που ήρθα με καθυστέρηση. Όσοι ενδιαφέρονται, η Αγγλία νίκησε τη Σλοβενία 1-0. θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι η επιδίωξη μιας αυτόνομης στρατηγικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 12 χρόνια είναι μια τεράστια σπατάλη και είναι κάτι το οποίο υποστηρίχθηκε παρόλα αυτά από το ΝΑΤΟ. Και ναι η Γαλλία έχει επανέλθει πλήρως στις στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ, αλλά η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει αυτόνομα τις δικές της στρατιωτικές ικανότητες είναι μια πάρα πολύ μακρινή λογική. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε λογικοί και να εμείνουμε θα έλεγα σε θέματα συμπληρωματικότητας, εξειδίκευσης με το ΝΑΤΟ να ειδικεύεται στις στρατιωτικές αποστολές. Και εδώ υπάρχει και χώρος για περαιτέρω ε, αγγλιογαλλική συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί ε, γενικότερα με ε, πολιτικές θα έλεγα δυνατότητες παρέμβασης. Έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική κατανομή εργασίας θα έλεγα η οποία θα βελτιώσει την συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας. Στην ουσία περιγράφουμε εκ νέου θα έλεγα με διαφορετικό τρόπο αυτό που ονομάζαμε στο παρελθόν Hearts and Minds. Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια μικρά σχόλια, αλλά θα ήθελα να θέσω και ορισμένες ερωτήσεις. Ίσως να καλύφθηκαν οι ερωτήσεις μου από κάποιους άλλους όσο ήμουν απόν. Αλλά η έκθεσή σας πώς έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται σήμερα η έκθεση αυτή της ομάδας Albright. Πιστεύετε ότι περιλαμβάνει ορισμένες παρατηρήσεις και νοτόμες, ρηξικέλευθες, ριζοσπαστικές. Δεν τις είδα εγώ με μια πρώτη ανάγνωση, διαρωτώ με όμως αν κάποιοι άλλοι έχουν καταλήξει κάπου. Θα ήθελα επίσης να μάθω πώς μπορούμε να τύχουμε περισσότερης υποστήριξης ευελιξίας και ε, σε εισαγωγικά επενδύσεων από πλευράς των Ευρωπαίων συμμάχων για τις λειτουργίες του ΝΑΤΟ και τις αποστολές του ΝΑΤΟ ιδιαίτερα στο Αφγανιστάν. Ξέρω ότι πολλές χώρες συμμετέχουν ευρύτατα στο Αφγανιστάν, όχι μόνο Αμερικανοί και Βρετανοί, το αναγνωρίζω. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια κάποια έλλειψη ευελιξίας και μια έλλειψη θα έλεγα ολόψυχη συμμετοχής κάποιων από τους Ευρωπαίους συμμάχους ε, στην προσπάθεια του ΝΑΤΟ. Και τέλος, και αυτό συνδέεται με το προηγούμενο, υπάρχει μια κάποια δυσθυμία γύρω από αυτό και πώς θα πρέπει να ανοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινή γνώμη στο ΝΑΤΟ. Οι λαοί μας έχουν αρχίσει και νιώθουν μια κάποια σύγχυση από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού θα έλεγα αυτών των δομών, των οργάνων, των συμμαχιών, υπάρχουν απλές λύσεις. Ξέρουμε τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία 12 χρόνια και οι οποίες δεν βοήθησαν ιδιαίτερα. Πρέπει να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να κάνουμε τη δουλειά που καλούμεθα να κάνουμε αποτελεσματικά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Υπάρχουν δύο όργανα στην ίδια πόλη που συναντιόνται και συνεδριάζουν, πολλές φορές για το ίδιο πράγμα. Αλλά πολλές φορές οι Ηνωμένε Πολιτείε λείπουν από κάποιες από τις σημαντικές αυτές συζητήσεις. Θα έπρεπε να το ξεπεράσουμε αυτό και να λειτουργήσουμε θα έλεγα πιο λογικά και να παράγουμε αποτέλεσμα το οποίο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του λαού μας. Ευχαριστώ. Μιλήσαμε πολύ για φιλοσοφία, αλλά νομίζω ότι με τη φιλοσοφία δεν θα προχωρήσουμε μπροστά σε αυτά τα τεχνικά θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια οικονομικά στοιχεία ένα πράγμα θέλω να θίξω. Αν όντως καταλήξουμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να συνδεθούν περισσότερο η μία με το άλλο, τότε αυτό σημαίνει ότι και η στρατηγική αλλαγή του ΝΑΤΟ θα πρέπει να υπάρξει και αυτή θα έχει επίσης μεγάλη επιρροή στην οργάνωση και στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρώ ότι ως βουλευτές πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας αυτό έχει να κάνει και με τη δημοκρατική πτυχή της οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ερώτημα ως προς αυτό. Είπατε στην αρχή της ομιλίας σας ότι στο ΝΑΤΟ αυτή η αρχή της συνένεσης κυριαρχεί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ε, μέτρο για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ. Αλλά εγώ έχω διαβάσει ότι γίνονται κάποιες σκέψεις από τον κύριο Ράσμουσεν αυτή η, αυτή η αρχή να ε, μεταφερθεί και σε άλλους τομείς. Αν αυτό μεταφερθεί και στα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά θα άλλαζε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ε, υπάρχει περίπτωση να αποδυναμωθεί ας πούμε η αρχή αυτή, ε, οι επιτροπές θα μπορούν ε, να αλλάξει η σύνθεσή τους. Αυτό θα σήμαινε, τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι θα υπάρξει μεγάλη αποκέντρωση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Και άλλο ένα ερώτημα. Ποιοι τομείς είναι αυτοί που θα ψηφίζουν με ενισχυμένη πλειοψηφία και αυτή η αρχή θα, είναι, θα ισχύει ας πούμε μία, ένα κράτος μία ψήφος και αυτό θα ισχύει και για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα λαμβάνονται υπόψη και τα μεγέθη των πληθυσμών των χωρών δηλαδή θα υπάρχει μια ιεράρχηση των, των μεγεθών αυτό θα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον να το δούμε ε, ας πούμε για τις μικρότερες κυρίως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο ένα ερώτημα γιατί ακούστηκε ότι δεν θα πρέπει να μιλούμε για το τι θα γίνεται με, τις, ε, με, τους, ε, με τα συστήματα άμυνας κτλ. Ε, ναι, αλλά το κόστος που υπάρχει για τις ευρωπαϊκές χώρες που θα τα φιλοξενήσουν Ήδη η Γερμανία και άλλες χώρες έχουν ε, συμφωνήσει για να υπάρξει αυτό το οπλικό σύστημα άμυνας σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Ο κύριος Ράσμουσεν μιλάει επίσης για, για σχέδια τα οποία θα κοστίσουν λιγότερο από 200.000 ευρώ. Από τον Πίτερ Φλόρι ε, διαβάζω, όταν ήταν και αυτός τότε ε, βοηθός του Γενικού Γραμματέα, ότι θα υπάρχει ένα σύστημα χωρίς εγκατάσταση τέτοιων ε, συστημάτων άμυνας, το οποίο θα, θα κόστιζε 100.000 ευρώ. Ένα σύστημα δηλαδή μόνο με μία εγκατάσταση, το ελάχιστο που σκεφτόταν τότε θα κόστιζε, έλεγε, 6 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δεδομένα λοιπόν του κυρίου Ράσμουσεν δεν είναι πολύ χαμηλά, δεν παρακλίνουν πάρα πολύ από αυτό. Δηλαδή δεν παρεκκλίνουν πολύ από, από την πραγματικότητα. Και κλείνοντας, μια παρατήρηση που σχετίζεται με αυτά που έλεγα και πιο πριν. Το συζητούσαμε και χτες και ο κύριο Σι νομίζω ήταν, ήσασταν εκεί. Ε, δεν θα πρέπει να το δούμε πολύ στενά αυτό το άρθρο για τον ΝΑΤΟ. Η ερμηνεία του άρθρου 5 είναι σημαντική. Και αν αρχίσουμε τώρα να δίνουμε διαφορετικές ερμηνείες, μπορεί όντως να υπάρξουν τεράστιες συνέπειες στο τι θα γίνει στο μέλλον γιατί μιλήσατε και για ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Ας πούμε, αν η προμήθεια πετρελαίου θα, θα ενέπιπτε σε δραστηριότητες του άρθρου 5. Αν ας πούμε υπάρξει μία επίθεση ε, σε ένα κράτος μέλος, αυτό επίσης εμπίπτει στο ε, άρθρο 5 και είναι της ίδιας σημασίας με την προηγούμενη επίθεση. Θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας για, μια προ... για έναν πρώτο γύρο απαντήσεων. Η Πασκάλ καταρχάς επειδή θα πρέπει να φύγει στις 7. Ευχαριστώ. Δεν θα απαντήσω σε όλα. Μπορούμε να έχουμε κατανομή αρμοδιοτήτων. Όσον αφορά τις ε, δυνατότητες της πολιτικές η γαλλική απάντηση είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αποκτήσει πολιτικές δυνατότητες που θα επικαλύπτονται με αυτές άλλων οργανισμών. Γι' αυτό τονίζουμε τόσο τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με άλλους οργανισμούς. Και εδώ περνάω και στην ερώτηση του κυρίου Βαν Όρντεν και υποθέτω ότι δεν θα σας εκπλήξει η απάντησή μου μιλήσατε για εξειδίκευση. Όντως αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες και αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε τρόπους συμπληρωματικής, παραπληρωματικής δράσης. Όμως δεν νομίζω ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε. Αν έχουμε μόνο στον ΝΑΤΟ στρατιωτικές δυνάμεις, σκληρή ισχύ και μόνο πολιτική δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι συμφωνώ με αυτό. Και επίσης, ε, από ό,τι κατάλαβα, έχετε κάποιες ε, ερωτήσεις ή αμφιβολίες για την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτόνομη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας πάντα είχαμε αυτή τη συζήτηση στις συνθήκες για και λέγαμε πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει μόνο όπου δεν παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Σήμερα έχουμε πολλά παραδείγματα όπου παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το ΝΑΤΟ και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας από το ΝΑΤΟ. Και ακόμα όσον αφορά την ε, περιβαλλική άμυνα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων αναφέρεται ως ε, βασική απαστολή η αντιπυραυλική άμυνα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πρόκειται για πρώιμη διαπίστωση. Είναι ένα θέμα και πολιτικό και οικονομικό και θα χρειαστούμε λίγο χρόνο στην σύνοδο της Λισαβόνας για να δούμε τι ακριβώς θα κάνει το ΝΑΤΟ. Και όπως είπε και η κυρία Λέζιν, κυκλοφορούν διάφορα νούμερα, άκουσα εδώ 200 εκατομμύρια ευρώ, να σας πω ότι στην τελευταία σύνοδο των Υπουργών ο Γάλλος Υπουργός είχε αμφιβολίες για αυτό το νούμερο και ήθελε να μάθει ποιο θα είναι το νούμερο. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητηθούν στο θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας. Εκτός μικροφώνου τα υπόλοιπα σχόλια. Ε. Πολύ σύντομα μια διευκρίνηση. Είπατε ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να έχει πολιτικές δυνατότητες που να βασίζονται σε άλλους οργανισμούς. Δέχεστε και το αντίστροφο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να έχει στρατιωτικές δυνατότητες που να βασίζονται σε άλλους οργανισμούς. Γιατί αυτό λέω. Όχι. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ένα σχόλιο για την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρέσβης. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με δύο πράγματα διαφορετικής φύσης. Από τη μία πλευρά έχουμε τον ατομο μια πολιτικοστρατιωτική οργάνωση η οποία λειτουργεί και στρατιωτικά. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ολοκληρωμένη ένωση, ένας ολοκληρωμένος οργανισμός. Βεβαίως έχει πολιτικές δυνατότητες, αλλά πρέπει να έχει και στρατιωτικές. Για μένα αυτό είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε στρατιωτικές δυνατότητες, Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε αλλού τη συζήτηση. Ποιος θα συνεχίσει. Λίγα σχόλια για τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Κοιτάξτε, τα στρατεύματά μας επιτόπου στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία Αργοζοβίνη, στο Κωσυφοπαίδιο, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε νατοϊκή αποστολή σε άλλες περιπτώσεις αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί τόπου η συνεργασία είναι πολύ καλή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια εδώ στις Βρυξέλλες. Και αν το κατορθώσουμε αυτό, η συνεργασία στο πεδίο της των επιχειρήσεων θα είναι ακόμη καλύτερη. Ένα από τα βασικά προβλήματα εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και η συμμετοχή ορισμένων μελών του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον οργανισμό. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό εδώ. Και κάτι τέτοιο θα ήταν ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός που θα μπορούσε να μας βοηθήσει και αλλού. Εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος όσο ο κύριος Βόλσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ. Πριν από δύο εβδομάδες ε, μας επισκέφθηκε η κυρία Άστον. Ο Ράσμουσεν ε, πήγε και στην ε, Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Ισπανία. Μικρά βήματα, όχι αρκετά, αλλά υπάρχει μια καλή κατεύθυνση και πρέπει να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα σχόλιο για την αντιπυραυλική άμυνα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Νομίζω ότι υπάρχουν παρανοήσεις εδώ αυτό που συζητάμε τώρα στο ΝΑΤΟ είναι να συνθέσουμε κάποια προγράμματα που ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ. Και αυτή τη στιγμή ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν πολύ καλή αντιπυραυλική άμυνα. Για παράδειγμα η Γερμανία. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί θέλουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύστημα και πρόκειται να πληρώσουν για αυτό. Τα 200 εκατομμύρια για τα οποία μιλάμε είναι το κόστος σύνδεσης των υπαρχόντων συστημάτων γερμανικού, το μελλοντικού, αμερικανικού, προκειμένου κατά αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε την προστασία των πολιτών μας. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να προστατεύουμε τα στρατεύματά μας, όμως εμείς ως πολιτικοί και μέλη αυτού του οργανισμού θέλουμε να παρέχουμε προστασία στους πολίτες μας. Συμφωνώ με την Πασκάλ ότι στη Λισαβόνα μάλλον θα ληφθεί κάποια απόφαση για το τι θα γίνει επ' αυτού και ποιο θα είναι τελικά το κόστος. Αυτή τη στιγμή καταλήγουμε στα τελικά συμπεράσματα και μιλάμε για 200 εκατομμύρια ευρώ εντός 10 ετών. Δεν είναι γιγαντιαίο ποσό και μιλάμε για σύνδεση με το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικό το οποίο οικοδομείται. Όσον αφορά τη συνένεση, υπάρχουν κάποιες γνώμεις ότι δεν πρέπει να ζητείτε συνένεση σε ορισμένα κομμάτια του ΝΑΤΟ. Όμως θεωρώ ότι το σύστημα λειτουργεί καλά και δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε. Και τίθεται και το ερώτημα του τι θα γίνει αν δεν απαιτείται η συνένεση στις επιτροπές. Τότε τα θέματα των επιτροπών θα καταλήγουν στον ΑΚ και τελικά η Πασκάλ θα είναι αυτή που θα πρέπει να βρει τη λύση. Και όσον αφορά το άρθρο 5, δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στην ερμηνεία του. Τώρα, για το άρθρο 4 που επίσης αναφέρθηκε και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Είναι ένα, νέο άνοιγμα το οποίο προτείνουν οι εμπειρογνώμονες αυτό και θα έπρεπε να το εξετάσουμε. Πολλά από τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί, οπότε θα απαντήσω όσα δεν απαντήθηκαν. Και θα κάνω και κάποια σχόλια γενικά. Καταρχήν, για τα θέματα τα πυρηνικά. Φυσικά είναι δύσκολα ζητήματα που πάντα είναι αντιφατικά πυρηνικά όπλα. Από τότε που εφευρέθηκαν πάντα ήταν αντιφατικό θέμα. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε επί τη βάση κάποιων βασικών αρχών. Καταρχήν, η αποτροπή των ε, πυρηνικών, ε, τέτοιων ε, επιθέσεων με πυρηνικά όπλα, η εξασφάλιση της ασφάλειας. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε βασικές αλλαγές, πρέπει να το κάνουμε προς το συμφέρον όσων πλήττονται. Και ούτως ή άλλως είμαστε μεταξύ συμμάχων θα γίνει αυτό. Και τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι και οι Υπουργοί Εξωτερικών ότι δεν θα υπάρχουν μεμονωμένα βήματα, θα υπάρξει συνένεση για να αναλυθεί οποιαδήποτε δράση. Δεύτερον, στο παρελθόν είχαμε μειώσει πολύ σημαντικά τον πυρηνικό μας οπλισμό. Το 80 υπήρχαν 7.000 πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη, τακτικά πυρηνικά όπλα, μικρό ο αριθμό δηλαδή. Τώρα έχουν μοιραστεί σε διάφορε χώρε, έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά όταν παίρνουμε, αποσύρουμε αυτά τα όπλα, αποσύραμε και άλλα ταυτόχρονα. Ας πούμε είχαμε την συνθήκη INF το 97. Οπότε το ερώτημα είναι, δεδομένου του ότι η Ρωσία, παρόλο που δεν είναι απειλή στο ΝΑΤΟ, αλλά η Ρωσία παρόλα αυτά έχει τεράστια όγκο πυρηνικών όπλων. Αν όμως πρέπει να κινηθούμε προς κάτι προς το μέλλον, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτή την πιθανότητα. Να υπάρχει δηλαδή ένας έλεγχος που θα ωφελεί τους πάντες των πυρηνικών όπλων. Και κάτι άλλο που είναι νομίζω σημαντικό. Φυσικά θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε σε έναν κόσμο όπου αν τα πυρηνικά όπλα δεν μπορούν να ε, σταματήσουν να υπάρχουν άμεσα, τουλάχιστον δεν θα παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι ένα. Αλλά απ' την άλλη, στο εγγύς μέλλον όλο και περισσότερες χώρες κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτήσουν δυναμι, δυναμι, δυνατότητες πυρηνικές. Οπότε Όλο και περισσότερες ε, ε, χώρες θα έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Αρκετές χώρες που ήδη προσπαθούν ε, έχουν, που, να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο ήδη έχουν δείξει ότι έχουν περίπου βαλιστικούς πυράβλους που, που ξεπερνούν τα πολύ κοντινά του σύνορα. Είναι διεπηρωτικοί. Οπότε Πώς θα βρούμε ένα ε, αντιστάθμισμα που θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα επιτεθεί κανένα στον ΝΑΤΟ. Πώς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό. Αν το καταφέρουμε θα είμαστε ε, οι πιο αποτελεσματικοί. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είναι ενισχύοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ στις ε, συζητήσεις για τον αφοπλισμό, τον πυρηνικό αφοπλισμό. Γιατί πυρηνικά όπλα θα υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα. Αν αύριο το ΝΑΤΟ, ας πούμε, ε, αποσύρει όλα του τα όπλα, θεωρείτε ότι αυτό θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας ε, που θα επηρεάσει και τη συμπεριφορά των υπολείπων χωρών ή θα είναι αυτό το αποφασιστικό βήμα που θα οδηγήσει όλους να αποσύρουν τα όπλα τους. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει η ε, συνθήκη για την μη διάδοση, οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει, ο πρόεδρος Ομπάμα επίσης κάνει πολλά σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Υπάρχουν και οι ε, ιδέες, οι απόψεις της ε, IAEA. E ε, είμαστε λοιπόν αρκετά πιο αποτελεσματικοί. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν λέω ποτέ, αλλά ό,τι είναι να κάνουμε, ας το κάνουμε ώστε να επιτύχουμε τους στόχους ασφαλείας. Ας μην είναι απλώς μια συμβολική κίνηση που δεν θα έχει καμιά επίπτωση και καμία, κανένα αποτέλεσμα. Επίσης αυτό που είπε ο Τζέφρι αυτό που θα σου έλεγα, Τζέφρι, είναι ότι οι περισσότερε στρατηγικέ δυνατότητε μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρώπη είναι ε, κρατικέ. Είναι ελάχιστε αυτέ που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Οπότε συμφωνώ με την ε, κυρία Πρέσβη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αυτονομία, έχει τη δυνατότητα να κάνει τις ε, αποστολές τις στρατιωτικές και αυτό θα μεγαλώσει. Ε, αυτό είναι σε, ο του ΝΑΤΟ γιατί το ΝΑΤΟ μπορεί να πάει σε περιοχές που ούτε καν θα σκεφτόσασταν ότι δραστηριοποιείται και μπορούμε να καλύψουμε πολλές ε, αποστολές ε, ειρηνευτικές και να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαδικασίες. Αλλά το θέμα είναι, ειδικά και με την χρηματοπιστωτική κρίση, είναι θέμα συνοχής. Δηλαδή, τι υπάρχει, τι είναι διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο και στο ε, ΝΑΤΟ, και αυτό που έχει το ΝΑΤΟ με τον Berlin Συν, με το Βερολίνο μπορεί να είναι διαθέσιμο θεωρητικά και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή το θέμα να χρησιμοποιεί ο καθένα μόνο του τα όπλα που έχει. Θέλουμε μια συνολική προσέγγιση, θέλουμε μια συνέργεια. Θέλουμε να αποφύγουμε τι επικαλύψει, θέλουμε να αποφύγουμε τι επαναλήψει. Θέλουμε τα, τα προγράμματα μα να είναι συμπληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά, να μην δαπανώνται τα χρήματα έτσι για, την, για πλάκα. Όταν ένα οργανισμό ηγείται, μιας ας πούμε ανάπτυξης μιας δυνατότητας, ο άλλος μπορεί να αναλάβει έναν πιο πολύ υποστηρικτικό ρόλο αντί να κάνει την ίδια δουλειά και να, να, να υπάρχουν επικαλύψεις. Όταν πριν από λίγα χρόνια, μια δεκαετία ας πούμε, η, οι προπολογισμοί των ΗΠΑ και των, ε, Ευρωπαϊκής ήταν ίδιοι για την άμυνα, η, είπα τώρα δαπανούν 73% του συνόλου του προπολογισμού του ΝΑΤΟ για αμυντικούς σκοπούς. Ε, η Ευρώπη δεν αυξάνει την, ε, ε, τον προπολογισμό του στον αμυντικό, ενώ πολλές χώρες το κάνουν, παρόλο που υπάρχει οικονομική χρήση. Η ολοκλήρωση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι ζωτική σημασία, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, αλλά και για να διατηρήσει και τις σχέσεις της και να διατηρήσει το ενδιαφέρον, τον, Ευρωπαϊ... αησία που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, για την έκθεση. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια διαδικασία μεταρρύθμισης από το 99 Ξεκίνησε από το 67 βέβαια με την τότε έκθεση. Οπότε πάντα δεν είναι ότι ο, ο οργανισμό δεν έκανε τίποτα τα τελευταία 20 χρόνια. Απλώ ήταν διακοσμητικό και ξαφνικά ε, εμφανιστήκαμε και είπαμε Α, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, να, κάνουμε, να δουλέψουμε σκληρά. Όχι. Είναι μια δουλειά εξελικτική που γίνεται. Δεν είναι επαναστατική. Και νομίζω ότι η έκθεση τώρα το φανερώνει αυτό δεν είναι ότι αποτύχαμε και ξαφνικά πρέπει να επαναφεύρουμε τα πάντα. Τούτου λεχθέντος υπάρχουν κάποια θέματα κανθόδια. Ας πούμε, η κυρία Ολμπράιτ και η ομάδα της ε, προτείνουν μια ευρύ, ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ. Είπα ασφαλεία της ενέργειας, ε, διάδοση κτλ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο επιλεκτικοί όμως. Υπάρχουν κάποια για τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα. Δεύτερον, ο κανόνα τη συνένεση που το ανέφερε η κυρία. Ε, επίσης, ένα άλλο παράδειγμα. Στην έκθεση της κυρίας Ολμπράιντ δεν υπάρχουν πολλά για τις επιχειρήσεις. Και αυτό δείχνει και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε και στο Αφγανιστάν. Τούτου λεφθέντο όμω. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στο Αφγανιστάν, το ΝΑΤΟ δεν θα είναι σε θέση να γυρίσει την πλάτη του στη διαδικασία σταθεροποίηση ε, ε, εγκαθίδρυση τη ειρήνη. Ήδη υπάρχει μεγάλη ανάγκη να παρέμβει το ΝΑΤΟ. Παρά τι δυσκολίε λοιπόν στο Αφγανιστάν, η τελική στρατηγική νομίζω ότι ε, συνεχίζει να περιλαμβάνει τον, την παρουσία του ΝΑΤΟ εκεί. Δεν λέω ότι δεν θα ξανακάνουμε κάτι τέτοιο μετά το Αφγανιστάν τέλος, και άλλο ένα ερώτημα της κυρίας Λέζιν για τα άρθρα. Δεν λέω ότι θα πρέπει να επαναερμηνεύσουμε τα άρθρα. Λέω απλώς ότι στην έκθεση Albright οι διαδιβουλεύσεις οδήγησαν στο άρθρο 4 ή έγιναν για το άρθρο 4. Αν όμως δείτε το άρθρο 4 λέει ότι αυτό είναι μια απάντηση μιας ε, απειλής. Εγώ δεν θέλω να δούμε μόνο αυτό όμως, όταν δηλαδή υπάρχει ένα σύμμαχος ο οποίος θεωρεί ότι κάπου υπάρχει μια απειλή, αλλά θέλω να συνδέσουμε τις διαβουλεύσεις αυτές με τις επίγουσες καταστάσεις του άρθρου 4 και να κάνουμε αυτό που κάνουν οι σύμμαχοι σε καθημερινή δουλειά. Να ελέγχουμε δηλαδή τα πράγματα και να ε, κάνουμε διαπραγματεύσεις, να ερχόμαστε σε επαφή. Δεν μπορούμε δηλαδή να, οι διαβουλεύσει να σχετίζονται μόνο με ένα άρθρο οι διαβουλεύσεις όπως λέτε στα γερμανικά είναι το ελιξίριο της ζωής. Ένα θέμα μόνο. Πολλά ακούστηκαν για διάφορα, αλλά θα ήθελα να επανέλθω στην τελευταία ερώτηση. Τι αφήνει ανοιχτό η σχέση αυτή. Πρέπει να υπογραμμίσουμε σε ποιο βαθμό η έκθεση υπογραμμίζοντας τις επιλογές γύρω από τις οποίες θα οργανωθεί η συζήτηση για τη στρατηγική, θα μπορέσει να βοηθήσει διαρθρωτικά στη μεταρρύθμιση της ε, συμμαχίας. Η διαδικασία αυτή λέει ο Τζέιμι ότι είναι συνεχής εδώ και 20 χρόνια. Οι συζητήσεις που γίνονται για το μέγεθος της συμμαχίας και για την ποιότητα της συμμαχίας απασχολούν συνεχώς τους Υπουργούς Άμυνας, σαν παράδειγμα, που το συζήτησαν και πριν 8 μέρες. Γι' αυτό λοιπόν στη Λισαβόνα θα μιλήσουμε για μια στρατηγική αντίληψη αλλά και για τις βασικές αρχές οργάνωσης και τη μεθοδολογία της συμμαχίας αυτής. Έτσι θα έχουμε και τον οδικό χάρτη αλλά ταυτόχρονα και τις οδηγίες χρήσης θα έλεγα των βασικών αποφάσεων, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα χαρακτηρίσει στο μέλλον για το πώς θα λειτουργεί η μηχανή του ΝΑΤΟ και πώς θα αναδιοργανωθεί. Σύντομα, δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Γιατί έχουμε ένα άλλο θέμα να συζητήσουμε για 10 λεπτά, ένα τέταρτο, άνα σύντομα. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι σύντομη, λέει η κυρία Σάντσου. Και εγώ έχω νιώσει ε, μια κάποια δυστημία γιατί συστηματικά κάθομαι πίσω από το Ζιρινόφσκι όταν πηγαίνω στην κοινοβουλευτική συνέλευση. είναι σαφές ότι έχουν μια ανταγωνιστική αντίληψη σε σχέση με μας και γι' αυτό ακριβώς μέχρι τώρα δεν έχουμε μπορέσει να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα και δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο επίπεδο της Ρωσίας στις συναντήσεις που έχουμε μαζί τους. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές οργανώσεις οι οποίες δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικές αλλά πρέπει να είναι συμπληρωματικές. Και όπως και η κυρία Αντριανή, ε, το δικό μου ευρωπαϊκό σχέδιο περιλαμβάνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναιρεί κανένα μέσο το οποίο να της προσδίδει αυτονομία, όπως το στρατιωτικό μέσο. Αν αυτό θα το κάνει διαρθρωτικά ή συμπληρωματικά με τον Άτο, τόσο το καλύτερο. Αν πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, θα το κάνουμε μόνοι μας και σε πολλές περιπτώσεις έπρεπε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες το ΝΑΤΟ ήταν ανίκανο να κάνει. Ιδιαίτερα τώρα, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με, τις, ε, με τη χρηματοδότηση και τις δυνατότητες της στρατογικές. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά αν παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και αυτό απαιτεί να υπάρξουν αλλαγές και σε εμά αλλά και στους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ. Και δεν μιλάω για τα στρατηγία μόνο, μιλάω επίσης και για τα εθνικά status quo τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις και δεν φεύγουν εύκολα από τις νατοικές αυτές αντιλήψεις. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση και της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα. Κάποια πράγματα μέσα από το ΝΑΤΟ δεν τα μπορούμε να τα πετύχουμε. Πρέπει όμως συνδυάζοντας τις προσπάθειές μας και να βρούμε τη χρηματοδότηση έτσι ώστε οι ικανότητες μας οι στρατηγικές να είναι χρήσιμες για την Ένωση αλλά και για το ΝΑΤΟ. Για το πυρηνικό κομμάτι. Έχει υπάρξει κάποια μικρή πρόοδος σε σχέση με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων και σε σχέση με τις παραδοσιακές παλαιότερες αντιλήψεις για το ρόλο του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λυπάμαι, αλλά με την κίνηση του Ομπάμα που μιλάει για έναν κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά όπλα. και αυτό δεν αφορά τα τακτικά πυρηνικά όπλα, αφορά την καταπολέμηση των μεθόδων ή μάλλον την ενίσχυση των μεθόδων καταπολέμησης της διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια εμείς ουσιαστικά διατηρώντας την ίδια αρχιτεκτονική ε, θα έλεγα ότι ενισχύουμε τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Υπάρχουν αντιστάσεις λοιπόν από τα διαφορετικά έτσι παραδοσιακά establishment και στο ΝΑΤΟ και στην Ένωση. Πρέπει να ξεπεραστούν αυτά. Χρειάζεται να συνεισφέρει και, η, και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία για την βελτίωση κάποιων στρατιωτικών ικανοτήτων και απαιτούνται επενδύσεις, γι' αυτό απαιτούνται χρήματα. Γι' αυτό και τέλος να πω ότι οι διαβουλεύσεις παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα πρέπει επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να συνδέσουμε τον άτομο με την κοινή γνώμη, όπου και αν βρισκόμαστε, στην Εθνικά Κοινοβούλια ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι περισσότεροι από αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα της άμυνας του ΝΑΤΟ έχουν γενικά στις, στην κοινή μας γνώμη πολλές φορές μια πάρα πολύ κακή εικόνα. Ξέρω ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε εμπλακεί στην εισβολή στο Ιράκ, αλλά πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είναι οι ίδιοι. Και για το Αφγανιστάν, εγώ ε, λέγω πάντα ότι το Αφγανιστάν είναι μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή. Αλλά δεν θα πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν θα πετύχουμε τίποτα πουλώντας το Αφγανιστάν στην κοινή γνώμη. Χρειάζεται λοιπόν διαφορετική αντίληψη, συγκλίνουσα αντίληψη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και στην ΚΕΠΑ δηλαδή να το πω καλύτερα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάπως τα πράγματα. Τάραντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ ότι βιαζόμαστε, αλλά σας υπενθυμίζω βεβαίως ότι σήμερα και είναι και η μεγαλύτερη ημέρα στο βόρειο ημισφαίριο, άρα έχουμε χρόνο. Λοιπόν, η Εστονία είχε πόλεμο ανεξαρτησίας και με την Ρωσία και με τη Γερμανία, άρα είναι αιμονή μας η ασφάλεια. Είναι δύσκολο να πούμε πολλά πράγματα σε δέκα σελίδες. Στην έκθεση Albright είδα μόνο μία πρόταση για τις απειλές που μπορεί να υπάρχουν έναντι του ΝΑΤΟ. Και η ερώτηση προς τον κύριο Σέι είναι η εξής θα έχουμε την ε, Σύνοδο της Λισαβόνας και είχαμε και αυτή την ομάδα που κατέληξε στο έγγραφο. Από εκεί και πέρα όμως θα υπάρξει κάποιος ε, στρατιωτικός σχεδιασμός πολύ λεπτομερής ε, π.χ. για θέματα ενεργειακής ασφαλείας, τι θα κάνει δηλαδή το ΝΑΤΟ αν ο στρατηγικός μας εταίρος ε, κόψει την παροχή στην Λευκορωσία και αντιμετωπίσουμε και εμείς πρόβλημα. Επίσης, ε, γενικά σε σχέση και με τις κλιματικές αλλαγές, πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέι και μετά λίγες λέξεις από καθέναν από τους ομιλητές. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντως, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο εφαρμογής ε, της στρατηγικής. Με ρωτήσατε για τη στρατηγική ασφαλείας της Εστονίας και των χωρών της Βαλτικής. Εδώ έχουμε δύο πτυχές. Καταρχάς, οι κλασικές ε, στρατιωτικές απειλές. Θεωρούμε ότι είναι μικρή η πιθανότητα γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ειρήνη στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Παρόλα αυτά, μία επίθεση θα μπορούσε να είναι καταστροφική και πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Η ασφάλεια συνήθως βασίζεται σε τέτοιου είδους ε, σενάρια που μπορεί να είναι σχεδόν απίθανα, αλλά θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά αν συμβούν. Γι' αυτό αυτό που κάνουμε είναι εντοπίζουμε και διασφαλίζουμε τη χώρα σας ότι είναι μέλη της συμμαχίας και έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν ε, απειλή για κάποιον. Αυτό κάνουμε τα 60 χρόνια της ε, ιστορίας μας. Στις επιχειρήσεις μας στα Βαλκάνια και στα, στο Αφγανιστάν ήταν οι τελευταίες, είναι αλήθεια, τέτοιου είδους επιχειρήσεις επί τη βάση του άρθρου 5, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε αν συμβεί οτιδήποτε. Υπάρχει όμως και η δεύτερη πτυχή, οι μη συμβατικές απειλές. Εσείς αναφερθήκατε στην ενεργειακή ασφάλεια, την πιθανότητα διακοπής της παροχής ενέργειας. Προφανώς εδώ υπάρχουν πολλά σενάρια, ακόμη και εμπορικές διαφωνίες που δεν έχουν να κάνουν με πολιτική βούληση, επίσης θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνικά προβλήματα, στους αγωγούς για παράδειγμα. Και άρα η λύση δεν θα είναι απαραίτητα στρατιωτική. Το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει με την προστασία των πολύ σημαντικών υποδομών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υποδομές μας για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δομές μας, για παράδειγμα το Συμβούλιο Ρωσίας-ΝΑΤΟ, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με διπλωματικό τρόπο. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι εδώ τις απαντήσεις μπορεί να τις δώσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ΝΑΤΟ. Με το δίκτυο, το πλέγμα ενέργειας, με τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας που μπορεί να σχεδιάσει και τα λοιπά. Άρα, στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας δεν βλέπω τον ΝΑΤΟ στον κεντρικό φορέα. Αν και πρέπει να εξετάσουμε και αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά, αν μιλάμε για δαλάσια ασφάλεια, για την προστασία των ε, των δεξαμενοπλοίων στη θάλασσα, εκεί θα μπορούσε να παίξει σαφώς σημαντικότερο ρόλο το ΝΑΤΟ. Τέλος, όσον αφορά το σενάριο του άρθρου 5, δεν πρέπει να αδιαφορούμε για τον ε, έλεγχο των όπλων. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε το καθεστώς CFE αυτή την περίοδο στον ΝΑΤΟ, γιατί υπάρχουν πολλές εντάσεις στα σύνορα και αλλού και αυτά δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας, όπως ακριβώς και οι παραδοσιακές απειλές στην ασφάλεια. Ευχαριστώ. Δύο σημεία. Καταρχάς το θέμα το πυρηνικό. Τακτικά πυρηνικά όπλα είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για μας. Γιατί με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα έχουμε 2.000 ρωσικά όπλα από το Καλίνιγκραντ μέχρι τα σύνορα της Νορβηγίας. Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ένωσης, αλλά μοιραζόμαστε την απειλή αν θέλετε. Έχουν υπάρξει μάλιστα και κάποια ε, ατυχήματα στα πυρηνικά υποβρύχια των Ρώσων που μας έχουν ε, κάνει να ανησυχήσουμε γιατί τα όπλα αυτά είναι λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. και έχουμε από την άλλη 200 όπλα Αμερικανών, Άγγλων και Γάλλων από την άλλη πλευρά και υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους αριθμούς. Τίθεται λοιπόν ένα θέμα σε σχέση με την ασφάλεια και τη διαχείριση όλων αυτών των όπλων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα συζητήσουμε. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και θα θέλαμε αυτά τα 2.000 όπλα να πάνε λίγο πιο ανατολικά και να μην είναι κοντά στα σύνορά μας. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να εκδηλωθούμε πρώτοι θα έλεγα θα πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση για την κοινοβουλευτική συνέλευση. Το Νοέμβριο θα φιλοξενήσουμε την κοινοβουλευτική αυτή συνέλευση μία εβδομάδα πριν από τη συνάντηση κορυφής της Λισαβόνας. Αυτό θα γίνει στη Βαρσοβία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η αντιπροσωπεία σας να είναι παρούσα με σωστούς όρους στην Βαρσοβία. Και ακριβώς έχει μεγάλη σημασία η διακοινοβουλευτική αυτή συνέλευση γιατί έρχεται μία εβδομάδα πριν από τη συνάντηση κορυφής και η φωνή των βουλευτών θα ακουστεί. Να καλωσορίσετε λοιπόν στην Βαρσοβία. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, ευχαριστώ όλους τους παρόντες και τον Τζίμι Σέι και τον κύριο Μπυρό. θα παρατείνουμε τη συνεδρίαση κατά 10 λεπτά. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Ο Κριστιαν θα μας μιλήσει για τη συνεργασία πολιτικών και στρατηγικών δυνατοτήτων. Είναι μια έκθεση η οποία θα εξεταστεί το Σεπτέμβριο στην Αρμόδια Επιτροπή αλλά ήδη ο Κριστιαν μπορεί να μας παρουσιάσει, θέλετε, τα, τις πρώτες γραμμές. Μεγάλη πρόκληση αυτή. Να δούμε ποιε είναι οι πολιτικέ επαφέ. Πριν από δύο μέρε, το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, συμφώνησαν για μια γενική δομή για το μέλλον τη ε, Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων που αφορά και τις δυνατότητες και την ανάπτυξη της ε, πολιτικής ε, ε, και των πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων. Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε τρεις τομείς. Καταρχήν το κενό που υπάρχει στην ανάπτυξη της διαχείρισης που υπάρχει στις πολιτικές και στρατιωτικές δυνατότητες, στο πολιτικό συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και τρίτον την διαλειτουργικότητα των, του εξοπλισμού. Νομίζω ότι οι ελλείψεις που υπάρχουν ή τα κενά που υπάρχουν ε, θα συζητηθούν ε, με τους, ε, σύμφωνα και με τους στόχους του Ελσίνκη που είναι και αρκετά προφανείς. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ότι στα, στα πλαίσια του, των στόχων του Ελσίνκη θα δεσμεύσουν 100.000 στρατιώτες, 100 πλοία για την, άμεση, για την ομάδα άμεσης πρόσβασης για το, που είχε ήδη δημιουργηθεί από το 2000. Αυτό μέχρι τις πρόσφατες ανακοινώσεις που είχαμε από το Συμβούλιο. Τώρα, για τις επιχειρησιακές ομάδες δηλώθηκε ότι από το, ήδη από, τον ε, από την 1η Γενάρη του 2007, δύο δηλαδή ομάδες πάντα σε stand-by, ε, δυνατότητα ανάπτυξης μέσα σε 10 μέρες μετά από την ε, απόφαση για την έναρξη της επιχείρησης. Οι ομάδε αυτές ε, μέχρι στιγμής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ και το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε μια ομόφωνη απόφαση που χρειάζεται. Δεν υπάρχει λοιπόν σαφή ορισμό του πώ θα χρησιμοποιηθούν οι ομάδε αυτέ και δεν υπάρχουν και συγκεκριμένα επιχειρησιακά καθήκοντα για το πώ αυτέ οι ομάδε θα, θα συνδυαστούν με τι πολιτικέ αποστολέ. Τώρα για τα δημοσιονομικά. τα κράτη-μέλη ε, χρηματοδοτούν αυτέ τι ε, ε, αυτές τις αποστολές, ενώ οι πολιτικές αποστολές χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ο συσχετισμός. Δεν υπάρχει δηλαδή λύση πώς να, πώς να χρηματοδοτήσουμε το, τις ομάδες αυτές και να γίνουν λειτουργικές. Τώρα, ε, αντιμετώπιση των, πολιτικών, ή, ε, των κρίσεων με πολιτικές δυνάμεις. Ήδη από το Γκέτεμπορκ το 2001 το συζητούμε το θέμα αυτό και πρόσφατα το 2008 αναδιατυπώθηκε το κείμενο αυτό και λέει ότι θα δώσουμε 5.000 αστυνόμους για διεθνείς αποστολές για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων. 1.500 θα μπορούν να αναπτυχθούν σε 30 ε, ημέρες και θα πρέπει να είναι έτοιμοι και ε, προετοιμασμένοι για τέτοιες, για τέτοιες ε, αποστολές. Επίσης αποστολές με ομάδες 10 εμπειρογνωμόνων που θα μπορούν να αποσταλούν μέσα σε 3 με 7 ώρες στον τόπο της κρίσης. Οι παρεμβάσεις λοιπόν και οι σχετικές ομάδες είναι κάτι που συνεχίζεται. Είναι δραστηριότητες ε, εν εξελίξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό προσωπικό που είναι διαθέσιμο είναι 11.000 πολιτικοί υπάλληλοι και τα κράτη-μέλη δεν έχουν, ε, ε, δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε καν 300 σε όλες αυτές τις αποστολές. Οπότε το κενό είναι μεγάλο και θα πρέπει να ορίσουμε και να τονίσουμε την ε, έλλειψη προσωπικού στους περισσο... στις περισσότερες αποστολές της ΚΕΠΑ και θα πρέπει να ενισχύσουμε την, ε, τις ε, δυνατότητες που έχουμε επαφών, λογισμικού, κατάρτισης, διαλειτουργικότητας κτλ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω επακριβώς τα, τους στόχους ε, που θα πρέπει να θέσουν τα κράτη-μέλη. Θα σας υποβάλω την έκθεση το Σεπτέμβρη. Αν τώρα πάμε στο συντονισμό ε, πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, ε, μιλούμε ότι για την ανάγκη της, του ορισμού των καθηκόντων, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουν στον αγώνα, αν μπορώ να το πω έτσι. Και ίσως θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κομισιόν και ε, Συμβουλίου. Είμαστε οι πρώτοι που αναλαμβάνουν, οπότε εγώ θα πρότεινα να δούμε το τι γίνεται με τα κεντρικά γραφεία, τα μόνιμα κεντρικά γραφεία, αν μπορούμε να έχουμε δηλαδή μόνιμα κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων, αν μπορεί να υπάρξει δια, λειτουργικότητα και για τις αστυνομικές και για τις στρατιωτικές και για τις πολιτικές αποστολές. Γι' αυτό θα χρειάζεται ένα κεντρικό γραφείο για να, για να συντονίζονται όλες αυτές οι ομάδες, να συντονίζεται και η ομάδα της, ε, από την Κομισιόν για την αντιμετώπιση κρίσεων και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις από μένα γι' αυτό. Επίσης, αν καταλήξουμε τώρα στο, στον εξοπλισμό, μιλούμε για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις, ας πούμε, ε, που θα έχουν τον ε, εξοπλισμό, θα πρέπει να υπάρχει απόθεμα για τις στρατιωτικές αποστολές και για τις πολιτικές αποστολές, επιχειρήσεις. Πώς ορίζουμε αυτό που χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς ε, οργανώνουμε ένα κοινό, την ύπαρξη κοινού εξοπλισμού και διαλειτουργικότητας αυτού, Γιατί αν έχουμε ένα πλαίσιο ας πούμε, επιχειρήσεων για τρία χρόνια, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή των κρατών μέλων, πρέπει να αλλάξουν, θα υπάρξει αλλαγή μονάδων. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα μόνιμο, μια μόνιμη μονάδα εξοπλισμού και πώς αυτό μπορεί να συνδυαστεί μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ε, δραστηριοτήτων. Γιατί σε τέτοια, ε, τέτοιος εξοπλισμό υπάρχει σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά δεν υπάρχει σε ένα ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Και αυτό σχετίζεται και με την οργάνωση της υπηρεσίας σχετίζεται και με θέματα προπολογισμού που επίσης πρέπει να λυθούν. Σχετίζεται και με το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, θα εφαρμόσουν αυτά που έχουν ε, αποφασιστεί. Υπάρχει μεγάλο κενό εκεί, μεγάλη έλλειψη. Και ο ΙΕ ή η ΙΠΑ μπορεί να έρθουν τώρα στις ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μα πούνε υπάρχει μια δεύτερη IT. Μπορείτε να βοηθήσετε. Εμεί, αν μα ρωτούσαν τώρα θα λέγαμε όχι, δεν μπορούμε να, το αναλάβουμε. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ευχαριστώ. Για τη δομή αυτή τη υπηρεσία. Πολλέ φορέ έχω μιλήσει. Πολύ σύντομα να πω και έξω ονόματος της ΓΚΟΕ ότι αυτή τη σύνθεση των, πολιτικών και στρατιωτικών ε, ε, επιχειρήσεων την αρνούμαστε υπό την ε, αιγίδα των, της υπηρεσίας. Η συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε κάνει και ακρόαση εδώ στην Επιτροπή, όπου δυστυχώς μόνο ένας, ένας υπήρχε ο οποίος είπε ότι ε, ο που εκπροσώπησε την πολιτική πτυχή αυτής της ε, συνεργασίας, ε, μια κυρία από τον Ερυθρό Σταυρό μάλιστα, και μας προειδοποίησε ότι περιορίζονται πάρα πολύ οι αρμοδιότητές της. Και ήταν πάρα πολύ λίγοι λοιπόν οι παρόντες εκείνη την ακρόαση. Είχαμε μια μια εκπρόσωπο από την κοινωνία των πολιτών που μας είπε ότι η συνεργασία αυτή θα αποτελούσε ίσως σημαντικό ρόλο για τις ε, υπηρεσίε ή για τις δραστηριότητες ε, για την, για την προστασία της κοινωνίας των πολιτών και αυτό ε, δυσκολεύει πάρα πολύ τη δική της ε, δουλειά, ε, γιατί πραγματικά πλήττεται η εξοπιστία των ε, υπηρεσιών αυτών ως ανεξάρτητων και ανθρωπιστικών υπηρεσιών. γιατί θεωρούνται ότι αυτοί οι στόχοι είναι ξαφνικά πολύ νόμιμοι και θεμητοί. Ε, αυτή ήταν η εμπειρία που είχαμε από, την, ε, από την ακρόαση. Έχουμε ακούσει παρόμοια σχόλια από πολλές τέτοιες οργανώσεις. Νομίζω ότι η, αρχή, η συνεργασία πολιτικών και στρατιωτικών επιχείρησεων δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να μας οδηγεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριος Γκουαλτιέρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χέλλερ για τις πληροφορίες που έδωσε. Νομίζω ότι ουσιαστικά δείχνουν ότι προετοιμάζει μια έκθεση φιλόδοξη αλλά και απαραίτητη γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σημερίζομαι λοιπόν τις θέσεις και το σχέδιο, τη δομή της εκθέσεώς του, η οποία μου φαίνεται ιδιαίτερα πιστική και ξεκινάει από μια, θα έλεγα μερικές φορές, ανησυχητική ε, πραγματικότητα και φυσικά και των στόχων που μπορεί να, να έχει κανείς έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες και χωρίς να αποκρύβει και την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να καλυφθούν δύο βασικά προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας για, την, για τον καλό συνδυασμό αν θέλετε των δύο διαφορετικών αυτών τρόπων αντιμετώπισης των κρίσεων στην εξωτερική διάσταση. Το πρώτο πρόβλημα είναι η αντίφαση ανάμεσα στην συνεχή εναλλαγή που υπάρχει και την ανάγκη από την άλλη για μόνιμες δομές και το άλλο πρόβλημα, η άλλη αντίφαση είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες δίδονται από τα κράτη-μέλη και οι χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και σε επίπεδο πολιτικών παρεμβάσεων και σε επίπεδο στρατηγικών παρεμβάσεων ξέρετε ότι υπάρχει ο μηχανισμό, υπάρχουν μηχανισμοί πάρα πολύ περίπλοκοι με φοβερούς συνδυασμούς. Τίθεται λοιπόν το θέμα της αντιμετώπισης του θέματος αυτού ε, με συνολικό τρόπο δημοσιονομικά για τη διαχείριση των κρίσεων επιμένω πάντα. Φυσικά η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι μια ενωτική θα έλεγα πλατφόρμα η οποία θα μπορέσει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα για να αντιμετωπίσουμε με πιο σωστό τρόπο τον συνδυασμό των κοινοτικών δυνατοτήτων, των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών διοικητικών δομών γίνεται μια προσπάθεια η οποία θα βοηθηθεί νομίζω από την ε, νέα αυτή υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Υπάρχουν και οι δυνατότητες που έχουν ε, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ε, που ασχολούνται με τα προγράμματα σταθεροποίησης. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνει ένα περαιτέρω βήμα και προς την κατεύθυνση αυτή σε επίπεδο Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων και συνδυασμού των προσπαθειών αυτής της υπηρεσίας με τις στρατιωτικέ υπηρεσίες. Κανένας δεν μπορεί να πει σε αυτή τη φάση πώς θα συντονιστούν μεταξύ τους οι εντελώς διαφορετικές δομές που ε, συμμετέχουν στη διαδικασία διαχείρισης των κρίσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι οι θέσεις του κ. Χέλλερ είναι ενδιαφέρουσες, πιστικές, Περιμένουμε το τελικό κείμενο για να τις αξιολογήσουμε, αλλά νομίζω ότι από πλευράς της πολιτικής μου ομάδας θα υπάρξει μια επικοδομητική στάση, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο συνενετικό, που θα ενισχύσει και θα επιταχύνει μια τόσο σημαντική και ευαίσθητη προσπάθεια για το μέλλον της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Ευχαριστώ. I really want to Ευχαριστώ. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Έλλερ γιατί είναι πολύ δύσκολο το θέμα και σας ευχαριστούμε λοιπόν που ασχολείστε με αυτό το τόσο κρίσιμη σημασία θέμα για την ε, κοινή πολιτική που μιλάτε για την ευρωπαϊκή αυτονομία σε επίπεδο ασφαλείας. Θα αναφέρω τρία σημεία απλά για να τα έχουμε επιτάπητος. Αργότερα θα τα συζητήσουμε. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα για τις ε, μόνιμες δομές και θα ήθελα να ακούσω τις ιδέες σας σχετικά. Δεύτερον, την ιδέα σας ε, για τα διαλειτουργικά συστήματα και αναμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και τρίτον, για την οικονομική πτυχή. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι έχει περάσει η ώρα και δεν περιμένω να ακούσω τώρα συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά ελπίζω ότι κατά την παρουσίαση του κειμένου σας θα έχουμε μια καλή συζήτηση από αυτόν. Και δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε και τώρα βεβαίως. Να πω ότι... Ακούσαμε τα πρώτα πράγματα για τις ε, πολιτικές και στρατιωτικές δυνατότητες. Τα πρώτα πράγματα που ακούσαμε είναι λογικά και πολλοί έχουν τις δικές τους ιδέες για αυτό το νέο σχέδιο που μπορεί να μας προσφέρει πολλά, αλλά που πρέπει να το χτίσουμε πολύ προσεκτικά αν θέλουμε κάποια πρόοδο σε αυτούς τους σημαντικούς τομείς και θα ακούσετε και τις δικές μας γνώμες αργότερα. Θα απελευθερήσω τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, και, και σας ευχαριστώ που καθίσατε λίγο παραπάνω. Κριστιαν, και σας υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε στις 9 τον για το Σιρένα. Το πιο υψηλά ιστάμενο στρατιωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κριστιαν, παρακαλώ, για να συνοψίσεις τα αγγλικά. So, so basically my suggestion is um, what we did is